παρατήρηση. Εγκρίνω λοιπόν τα πρακτικά αυτά. Προτού τώρα περάσουμε στο πρώτο θέμα της απογευματινής μας ε, συζήτησης, θα ήθελα να πω ότι έχουμε στα θεωρία μια επίσημη αντιπροσωπεία από την Βουλή της Νοτιοαφρικής. Σας καλωσορίζω έχουν έρθει οι βουλευτές αυτές από την Νότιο Αφρική για να συμμετάσχουν στην 14η ε, μεικτή κοινοβουλευτική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ανεχειριστώ τον Ζωμαϊ Λουίς Φάπς που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για Εμπόριο. Συνοδεύεται από τον κύριο Τόμας Τέξη, πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και πέντε άλλοι βουλευτές της ε, Νοτιοαφρικής Βουλής. Ξέρετε ότι συμμερίζομαστε με την Νότια Αφρική τις ίδιες αρχές για τη δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και συνεργασία. Δεν είναι μόνο μια περιφερειακή δύναμη της Νότιας είναι και μια αναδυόμενη διεθνής δύναμη. και αντιμετωπίζουν και εκείνοι βέβαια τι προκλήσει από την διεθνή οικονομική κρίση. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε το διάλογο και να ενδυναμώσουμε τις σχέσει μας και τη συνεργασία μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όχι μόνο για να επιλύσουμε την τρέχουσα ε, κρίση και να βρούμε σωστές ε, στρατηγικές, αλλά να συνεργαστούμε και για να υπάρξει μια διεθνής ε, δομή διακυβέρνηση που θα μας ωφελήσει όλους. Σας καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να σας πω ότι μπορούμε τώρα να περάσουμε στην έκθεση Μπροκ για τις ε, θεσμικές πτυχές ε, της ε, ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.